Μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Οπότε ολοκληρώνονται οι ομιλίες και να απαντήσει τώρα ο Επίτροπος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι πιθανώς θα εγκριθεί το ψήφισμά σας για την Βοσνία Ζεγοβίνη και συγχαίρω τον κύριο Πρέντα γι' αυτό. Είναι υψηλού επίπεδου η έκθεσή του και ευχαριστώ και όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου που συμμετείχαν στην ε, εκπόνησή της και στη σημερινή συζήτηση και έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για την ε, ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Σημειώνουμε το ψήφισμα πολύ προσεκτικά και όλες τις απόψεις του Κοινοβουλίου συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εξεφράστησαν κατά τη σημερινή συζήτηση. Ιδιαίτερα συμμεριζόμεθα την άποψη του Κοινοβουλίου ότι οι αρχές που θα προκύψουν, που προέκυψαν συγγνώμη, τα αποτελέσματα των εκλογών του Οκτωβρίου 2018 πρέπει να οδηγήσουν σε σχηματισμό κυβέρνησης που θα βοηθήσει την προώθηση των σχέσεων ε, Ένωσης Βοσνίας Ζεγοβίνης. Και επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη και το κείμενο της Κομισιόν που ε, αναφέρει ότι το ενδεχόμενο πρότασης ε, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ως υποψηφίας χώρας θα εξαρτηθεί από τις απαντήσεις στο κείμενο. Επίσης, η λειτουργία της ε, Συμφωνίας ε, Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και της ε, κοινοβουλευτικής διάσκεψης είναι σημαντικά θέματα και θα τα, θα τα θίξω με την ηγεσία της Βοσνίας Αζεγοβίνης και θα αξιολογήσουμε την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης για να εκπονήσει την επόμενη γνώμη της από αυτόν. Επίσης, η Κομισιόν δεν θα αφιστεί προσπαθειών για να στηρίξει την Βοσνία Ζεγοβίνη στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η κυρία Μάλετιτς και άλλοι είπαν ότι πρέπει να εντοπίσουμε και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες μέσω προγραμμάτων. Συμφωνούμε, θα το κάνουμε. Και βεβαίως θα συνεχίσει η Κομισιόν να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για τις ενδεχόμενες εξελίξεις όσον αφορά τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Ο κύριος Τσάμπα έχει το λόγο, υπουργό. Παρακαλώ. Α, ευχαριστώ. Και εκ νέου επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω εκ νέου τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει και συνολικά το Κοινοβούλιο. Η Ρουμανία ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου έχει θέσει ως προτεραιότητα να είναι φίλη με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων βοηθώντας τις να προχωρήσουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είμαστε αποφασισμένοι να βοηθήσουμε όλες τις χώρες βεβαίως εφόσον υιοθετήσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και σε ό,τι αφορά τη Βοσνία Ζεγορμίνη υπάρχει επίγουσα ανάγκη διαμόρφωσης κυβέρνηση σε κάθε επίπεδο και ουσιαστικής εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Θα επισκεφθώ το Σαράγεβο και η Προεδρία μας θα επισκεφθεί όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ούτως ή άλλως πριν τις συζητήσεις, ε, τις κρίσιμες συζητήσεις του Συμβούλιο τον Ιούνιο. Ταυτόχρονα Μία από τις εκδηλώσεις της Προεδρίας είναι να μπορέσει η περιφέρεια να συμφιλειωθεί με το παρελθόν της με έμφαση ακριβώς στα Βαλκάνια και υπογραμμίζοντας τη σημασία να ξεπεράσουμε την ε, ρητορική του διχασμού και να υπάρξει μια πραγματική συμφιλίωση στην περιοχή. Ευχαριστώ και για την προσοχή σας. Ο εισηγητής τώρα, κύριος Πρέντα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ. Έκανα αυτή την υπόδειξη, μάλλον τη δέχτηκα, κύριε Τσάμπα. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να συνεργαζόμαστε με τους νέους, να τους μιλούμε για την Ευρώπη και να δούμε τι μπορεί να γίνει στα πλαίσια της συμφιλίωσης. Έχουμε έναν Βρετανό συνάδελφο, ο οποίος μίλησε για το Star Trek. Ο συνάδελφος, ο Έλληνας, μίλησε για το ΝΑΤΟ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ήθελα να τον ρωτήσω τότε γιατί τον Πειραιά δώσατε στους Κινέζους όταν μιλάμε για διακυβεύματα δηλαδή. Το θέμα όμως της ε, Βοσνίας Ερζεγοβίνης ε, εντάσσεται στα Δυτικά Βαλκάνια. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή χώρα. Το, 95% των Κροατών της Βοσνίας Ερζεγοβίνης είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Υπάρχουν ε, πολλές ε, εθνότητες που είναι πολύ πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και οι Κροάτες. Οι Κροάτες πρέπει να σκέφτονται και τους άλλους, όχι μόνο τον εαυτό τους. Ε, θα είναι υπέρ της ολοκλήρωσης και της προσχώρησης όταν σκεφτούν και τους άλλους, όχι μόνο τους ίδιους τους εαυτούς τους που είναι ήδη Ευρωπαίοι πολίτες. Θα πρέπει να εντάξουμε και τα πολιτικά κόμματα σε αυτό το δίκτυο. Δεν υπάρχουν φιλελεύθερα ε, κόμματα ή σοσιαλιστικό κόμμα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αν δεν έχετε επαφές ε, επιτόπου, τι μπορείτε να κάνετε. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά για να βοηθήσουμε την Βοσνία Ερζεγοβίνη να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να περάσουμε αυτή την στήρα ρητορική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον εισηγητή Πρέντα. Λίγη η συζήτηση, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Διακόπτουμε για δύο λεπτά και μετά θα αρχίσει η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.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 Κύριε Πρωθυπουργέ της Ιταλικής Δημοκρατίας, σας ευχαριστούμε πολύ γιατί δεχτήκατε την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μας εκθέσετε τη δική σας άποψη και όραμα για το μέλλον της Ευρώπης από πλευράς Ιταλικής Δημοκρατίας. Η Ιταλία είναι μία από τις ιδρυτικές χώρες και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί μπορούμε να προωθήσουμε αυτή τη συζήτηση για το μεγάλο αυτό ζήτημα που αφορά 500 εκατομμύρια κατοίκους. Υπάρχουν θέματα μεγάλου ενδιαφέροντος για τους Ευρωπαίους πολίτες. Εμείς θέλουμε να είμαστε η δημοκρατική καρδιά της Ευρώπης. Έχουμε εκλεγεί άμεσα από τους πολίτες και δώσαμε μεγάλη μάχη για την αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1,1 στο 1,3 όσον αφορά τους ίδιους πόρους. Ασχοληθήκαμε με το θέμα της μετανάστευσης. Είμαστε υπέρ περισσότερων επενδύσεων προς την Αφρική για να επιλύσουμε το ζήτημα από τη ρίζα του. Εγκρίναμε μία πρόταση που υπάρχει επιτάπητος σχετικά με αυτό το θέμα και θα θέλαμε και εμείς να συμμετάσχετε σε αυτή τη διαδικασία ως πρωταγωνιστής έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις χώρες προς νότον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πλήττονται ιδιαίτερα από το προσφυγικό. Ως προς το Brexit, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσεται υπέρ των πολιτών και της προστασίας τους που ζουν στις Βρυξέλλες. Ζητήσαμε μια ουσιαστική αύξηση πόρων έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαρθρώσεων να ταχθεί υπέρ της ανάπτυξης και ως προς την εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν τον προσωρινό πρόεδρο της ε, Βενεζουέλας, τον κύριο Γκουαϊντό. Ένα άλλο θέμα που ε, εντάσσεται στο πρόγραμμα της ε, κυβέρνησής σας επίσης, αφορά ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να μετράει περισσότερο μέσα στα πλαίσια του νομοθετικού του έργου και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Σας δίνω το λόγο για να μας πείτε τη σκέψη της Ιταλικής Δημοκρατίας για το μέλλον της Ευρώπης. Intanto vi potete registrare per il catch the eye con il Presidente del Consiglio ζητήσετε να καταχωρήσετε το όνομά σας για το Catch the Eye στο τέλος της παρέμβασης ε, του Ιταλού Πρωθυπουργού. Κύριε Πρόεδρε Ταγιάννη, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε Κατάινεν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι πραγματικά τιμή για μένα να απευθύνομαι σήμερα ενώπιόν σας και το λέω με ειλικρίνεια για να περιγράψω το μέλλον της Ευρώπης ε, σύμφωνα με τις θέσεις της Ιταλικής κυβερνήσεως. Η δέσμευση για το μέλλον της Ένωσης μας ξεκινά με μια πραγματικά συγκινητική αναφορά στον Αντώνιο Μεγαλίτσι, έναν Ιταλό που όριζε τον εαυτό του ως ερωτευμένο με την Ευρώπη, που ήταν θύμα των επιθέσεων πριν από δύο μήνες στο Στρασβούργο της τρομοκρατική βαρβαρότητας. Σε έναν παγκοσμιωμένο κόσμο όπου η οικονομία φαίνεται πως ε, πήρε τα πάνω της σε σχέση με, το, με, τα δικαιώματα και όπου η οικονομία απομακρύνεται ε, από τις θέσεις των πολιτών μας πρέπει να θέσουμε ερωτήματα για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρμοδιότητές της, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά κράτη, τα κράτη-μέλη, δηλαδή μόνα τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σύνθετες παγκόσμιες προκλήσεις. Το κοινό ευρωπαϊκό οικοδόμημα, πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι, περνά μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα φαίνεται ότι έχασε την ικανότητα να προχωρά η, συγκυρία, ιστορική συγκυρία που είναι πολύ σύνθετη είναι, αποτελεί μια πρόκληση για όλους μας ε, από τα διάφορα θεσμικά επίπεδα να αντιμετωπίσουμε εξαιρετικά κρίσιμα ζητήματα όπως έκαναν στο παρελθόν και άλλοι που μας προκάτοχή μας και εμείς τώρα καλούμεθα να καταβάλουμε μια κοινή προσπάθεια με πλήρη επίγνωση των ευθυνών μας. Έχουμε την ευθύνη να θέσουμε εκ νέου σε κίνηση το ευρωπαϊκό εγχείρημα επιτρέποντάς του να αποκτήσει αξιοπιστία και συνοχή για να αυξήσει την βιωσιμότητα, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητά του. Οι προκλήσεις σήμερα είναι νέες, σύνθετες, απαιτούν όραμα, και αν μου επιτρέπετε και μία δόση δημιουργικότητας. Προϋποθέτουν ωστόσο κατά βάση επίγνωση της αποστολής μας στον κόσμο. Τα μεγάλα αιτήματα που πρέπει, στα οποία πρέπει να δώσουμε απάντηση είναι ερωτήματα ουσίας. Ποια Ευρώπη θέλουμε. Ποια Ευρώπη χρειαζόμαστε. Πώς βλέπουμε εμάς στην Ευρώπη Αυτά είναι ερωτήματα που έχουν συνδυσιακό χαρακτήρα και απαιτούν μεγάλη, μεγάλη αυτεπίγνωση. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει εκλεγεί απευθεία από τους Ευρωπαίους πολίτες και που είναι αυθεντικός θεματοφύλακας της Ευρωπαϊκής Κυριαρχίας πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε και πρέπει να είμαστε ένας λαός ο ευρωπαϊκός λαός σε μια διαδικασία ενοποίησης που μας δημιούργησε μια κοινότητα πεπρωμένου πέραν οποιασδήποτε νομικής, ε, ε, νομικής αναγνώρισης. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα βίωσε σημαντικές στιγμές πρόοδου εδώ. Η ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης χαράχθηκε από βαθιές διαιρέσεις, από συγκρούσεις, από αντιπαραθέσεις που διαμόρφωσαν έναν, ε, ε, μια εθνική ταυτότητα, πλου, εθνικές ταυτότητες πλούσιες, ε, πολυ, πολυ, πολυγλωσσικές και που όμως λειτουργήσαν και θετικά νομικά και κοινωνικά. Ενσωματώσαμε στα οικονομικά μας συστήματα, τα εκπαιδευτικά μας ε, συστήματα, την, ε, την κοινωνική μας νομοθεσία, δίνοντας χώρο σε κυριαρχίες και πηγαίνοντας σταδιακά από το κράτος στην Ένωση. Επιτρέψαμε στα, στους πολίτες των κρατών μελών να κυκλοφορούν ελεύθερα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναν ενιαίο νομικό χώρο. Η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων πολύ περισσότερο και από την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και των ε, κεφαλαίων ήταν μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Σκεφτείτε ακριβώς το βάρος του, του εθνικιστικού μίσους που είχε πλήξει τον, την Ευρωπαϊκή Ήπειρο το πρώτο ήμιση του 20ου αιώνα και που σε δύο παγκόσμιους πολέμους. Οι Ευρωπαίοι, ιδίω οι νεότεροι, δεν θέλουν να εγκαταλείψουν αυτή την θεμελιώδη ελευθερία κίνησης, χάρη στη, στα οποία μπόρεσαν με τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν να αποκτήσουν πλούτο ε, πολιτισμικό ε, και εμπειρίες υιοθετώντα και ε, αντλώντας από διάφορες εθνικές εμπειρίες και από την ικανότητα να συμμετάσχουν σε, μια κοινή, σε ένα κοινό συνέστημα. Η διαδικασία δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού λαού ε, τροφοδοτήθηκε και, από τα νομικά εργαλεία καρπό μιας δια, πολιτισμικής διαδικασίας κοινή υιοθέτηση της μιας νομικής ταυτότητας, της δημιουργία ενός ίντεμ, ενό ε, ευρωπαϊκού δήμου. Το έργο στο πλαίσιο αυτό του, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ήταν καθοριστικός και για την εθνική συνταγματική διαμόρφωση. Μέσω αυτών δημιουργήθηκε ένας ευρωπαϊκός νομικός χώρος όπου μπορούσε να αναγνωρίσει τον εαυτό του πολίτης και να αναζητήσει προστασία μέσω ενός πλήρους ολοκληρωμένου συστήματος προστασία σε πολλά επίπεδα των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου που στηρίζεται σε μια κοινή παράδοση συνταγματικών ε, ταυτοτήτων. Το εξελιγμένο αυτό σύστημα δικαιοδοτικής προστασίας ε, που εντάσσεται πλέον ε, με ανεξίτηλο τρόπο στην κοινή νομική κληρονομιά της Ένωσης αποτελεί μια πολιτισμική κατάσταση που πρέπει να προστατεύσουμε ακριβώς λόγω των ενάρετων συνεπειών που επέτρεψαν να μπορέσει συλλογικά ο Ευρωπαίος πολίτης να έχει την επίγνωση της Ευρώπης τροφοδοτώντας την ε, κατανόησή του ότι μετέχει σε ένα κοινό έχειν μετέχει, ότι μετέχει σε έναν λαό που, μετέ, που περιλαμβάνει τα ίδια γόνιμα στοιχεία πολιτισμού. Παρόλα αυτά δεν καταφέραμε να γίνουμε ακόμα και πλήρως ένας λαός. Δεν είχαμε το θάρρος να οικοδομήσουμε ένα ε, ολοκληρωμένο μοντέλο που πέραν της ρητορική θα ενθάρρυνε την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δήμου. Ιδίως μετά το 1989 έλειψε με κάποιες εξαιρέσεις βέβαια μία ένα πραγματικά πολιτικό όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία προοπτική στο μακρύ χρόνο, με πρόβλεψη στο μέλλον. Γι' αυτό, χωρίς την οποία το όνειρο τελματώνει στην άμμο και χάνει τη δυνατότητα να προχωρήσει. Αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ιδρυτικών πατέρων της Ευρώπης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η... Το έλλειμμα, λόγω του ελλείμματος αυτού του οράματος των τελευταίων 30 ετών, η Ευρώπη περιορίστηκε στο στην οικονομική της διάσταση που οδήγησε σε μείωση της ε, ρυθμιστικής προσέγγισης σε κρίσιμους οικονομικούς τομείς, περιορισμό της κοινωνικής υποστήριξης και του, του, του κράτους πρόνοιας που αύξησαν συνολικά τις ανισότητες πλούτου και ανισότητες ευκαιριών. Ιδίω με την άφηξη της οικονομικής κρίσης, η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση υποστήριξε πολιτικές λιτότητας με στόχο αποκλειστικά να περιορίσουν τα, τα κρατικά ε, τα κρατικά χρέη και να κρατήσουν το ποσοστό πληθωρισμού του κοινού νομίσματος όσο χαμηλότερα γίνεται. Εις βάρος μερικές φορές και της κατανάλωσης με καταστροφικές συνέπειες σε κοινωνικό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή πολιτική ενώπιον αυτής της ε, οικονομικής κρίσης ε, φοβήθηκε την και έχασε σταδιακά την επαφή με τον λαό, καθιστώντας ολοένα και μεγαλύτερη την απόσταση, όχι μόνο γεωγραφικά, μεταξύ Βρυξελών και των περιφερειών της Υπήρου μας. Σταδιακά η πολιτική έχασε την νομιμοποιητική και αντιπροσωπευτική της διάσταση. Εμφανίζεται στους πολίτες ολιγαρχική και απόμακρη, αδύναμη να καταλάβει τις πραγματικές ανάγκες της ε, κοινωνίας. Έγινε, όπως σωστά το είπε η πολιτιολόγος Άννα Γελόνκα, μία τελετουργική παράμετρος κάλυψης παγκοσμιοποιημένων δραστηριοτήτων που εν γέννη είναι ακατανόητες και μυστικές. Η δυνατότητα άρνησης, η άρνηση που δείχνει ο ευρωπαϊκός λαός της ελίτ ε, απευθύνεται σε εμά, μας θυμίζει ότι η πολιτική που υποδουλώνεται στην οικονομία χάνει τις αρμοδιότητές της, χάνει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στα αιτήματα. Βρισκόμαστε σε μια στιγμή αποφασιστική για την ιστορία της Ευρώπης. Μας αναμένουν καθοριστικές αποφάσεις για το μέλλον μας. Ο ευρωπαϊκός λαός έχοντας ξαναεμφανίζεται στο προσκήνιο της ιστορίας και ζητά επιτέλους να τον ακούσουμε. Ζητά να υπάρξει μια αποφασιστική αλλαγή της μεθόδου και της προοπτικής. Είναι μια ευκαιρία, πολύτιμη θα έλεγα, να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο, να επενδύσουμε στην μείωση της, από, της απόστασης μεταξύ κυβερνώντων και κυβερνομένων που τροφοδοτήθηκε από τη σιωπή, την αδιαφορία και την προσπάθεια ελαχιστοκυπήσης του μεγέθους για να μειώσουμε την, ε, τον κίνδυνο εσωτερικής έκρηξης του κόσμου που βιώνουμε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την σύγκρουση. Πρέπει να είμαστε όμως σε να την διακυβερνήσουμε αυτή. Δεν πρέπει να από περιοριστούμε σε έναν στήρο συντηρητισμό που αρμόζει σε μια πολιοκυμένη πόλη. Αντίθετα, πρέπει να εκφράσουμε με νέες μορφές δημοκρατίας την ικανότητά της να καινοτομήσει αναλαμβάνοντας, αναλαμβάνοντας και τον κίνδυνο να εγκαταλείψουμε κάποιες ε, παρελθούσες βεβαιότητες, κάποια μοντέλα ανάπτυξης ή σχέσεις δυνάμεων που δεν ανταποκρίνονται πλέον με την πραγματικότητα. Δεν πρέπει να αφήνουμε κοινωνίες φτωχοποιημένες που εξαρτώνται από, αβέβαια, από ένα αβέβαιο μέλλον. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αμφισβήτηση και σε εξέγερση με απρόβλεπτες συνέπειες όπως βλέπουμε σε διάφορα φαινόμενα σε διάφορες χώρες της Ένωσης. Ο ευρωπαϊσμός του 21ου αιώνα, κατά την άποψή μου, προϋποθέτει αναπόφευκτα να ξανασκεφθούμε ριζικά τις μορφές και τους θεσμούς που χαρακτήρισαν την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης τα τελευταία 30 χρόνια. Απαιτούν επιγόντως μία αυθεντική σύγκληση που για κάποιους οδηγούν στο να επανέλθουμε στο αρχικό, στην αρχική εικόνα του ευρωπαϊκού οράματος. Η Ευρώπη που φανταζόμαστε θα πρέπει να είναι μια Ευρώπη που επιτρέπει να προχωρήσουμε, όχι μόνο που να σταθεροποιούμε, να σταθεροποιεί, ή προς όφελος των πολιτών. Η προς των αλλάζει γρήγορα. Οι νέες γεωπολιτικές ισορροπίες είναι εξαιρετικά ε, ασα, ασαφείς κάποιες δυνάμεις που δεν μπορούν να, να καταφέρουν να δημιουργήσουν πραγματικούς πόλους διεθνούς ε, επιρροής ε, αυξάνουν παρά τα αυτά την επίδρασή τους. Στο πλαίσιο αυτό κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να παίξει μόνο του έναν σημαντικό ρόλο. Εξού και η ευχή για μια ενωμένη Ευρώπη με θέση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτός είναι ένας δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε με συντονισμένο τρόπο, με μια φωνή. Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να μιλήσει στον κόσμο. Μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, φιλόδοξη, συνεκτική, είναι αναγκαία κατά βάση για να βελτιώσουμε την ικανότητά της να συνομιλεί με τις Ηνωμένε Πολιτείες, όπου ίσως είχα πει στην πρώτη παρέμβασή μου ε, στο Ιταλικό Κοινοβούλιο πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό στην συζήτηση με την Ουάσιγκτον για να διαφυλάξουμε το στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεών μας. Εδώ πρέπει να αναδείξουμε αυτά που μας ενώνουν βασικές αξίες και όχι τυχόν διαφορές και ελλείψεις κατανόησης. Ταυτόχρονα, μια ισχυρή Ευρώπη είναι αναγκαία για να μας επιτρέψει να συνεχίσουμε το διάλογο με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στην παγκόσμια σκηνή. Η Ρωσία και η Κίνα είναι μέρη οποιασδήποτε λύση στις βασικές παγκόσμιες κρίσεις, ακόμα και στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα κερδίσει αν αποποιηθεί της δυνατότητας να συνεχίσει το διάλογο με τη Ρωσία και την Κίνα ή να αποκτήσει ή να υποστηρίξει τις, απο, τις ε, απομονωτικές τους ε, προσεγγίσεις. Πώς θα γίνει όμως αυτή η ισχυρή Ευρώπη που όλοι θέλουμε. Πρέπει βέβαια να, να προχωρήσουμε στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής άμυνας χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες ε, που μας, παρέχει, που μας η ΠΕΣΚΟ, η διαθρωμένη μόνιμη συνεργασία, προς μία ευρωπαϊκή άμυνα που δεν είναι μόνο ε, που δεν δημιουργεί προβλήματα στη σχέση μας με, την, με τον ΝΑΤΟ αλλά αντίθετα είναι και ένα θετικό συμπλήρωμά του. Αυτό επιτρέπει και μεγαλύτερη ασφάλεια των, πολιτών, των πολιτών μας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να συνεχίσει να έχει στενούς δεσμούς στην άμυνα και την ασφάλεια με το Ηνωμένο Βασίλειο και μετά το Brexit. Βασική προϋπόθεση για μια ισχυρή Ευρώπη στον κόσμο είναι να εξασφαλίσουμε κατά βάση την αλληλεγγύη και τη συνοχή μέσω της συλλογικής ε, συνεργασίας των κρατών μελών. Η μετανάστευση και η οικονομική διακυβέρνηση είναι βασικοί πυλώνες για να υποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Οι αρχές αυτές δεν πρέπει να οδηγήσουν σε διαιρέσεις τα κράτη-μέλη. Αντίθετα, τα κράτη-μέλη πρέπει να έρθουν κοντά στα μεγάλα αυτά ζητήματα που πρέπει να είναι κομμάτια της ε, ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ακριβώς την αδυναμία της Ευρώπης να προτείνει να λειτουργούμε με τρόπο ίσο προς ίσο μεταξύ των πλευρών. Η, το θέμα της μετανάστευσης ήρθε αργά στην Ευρώπη και χάρη στην Ιταλία. Η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις ε, μεταναστευτικές ζωές ως μία επίγουσα ανάγκη, αλλά πρέπει να αποκτήσει μία σταθερή θέση με αποτελεσματικό τρόπο. Και απευθύνομαι σε εσά με μία έκκληση που την επαναλαμβάνω σε κάθε σύνοδο κορυφής και σε κάθε άτυπη συνάντηση στην οποία μετέχω. Δεν πρέπει να, να καθυστερήσουμε περισσότερο την υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου της 28 Ιουνίου πέρυσι. Χωρίς μια αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών δεν τηρείται καν η αρχή της Ενωμένης ΕΕ. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική που θα αντιμετωπίζει σωστά και με τη σωστή προτεραιότητα τις πρωτογενείς μετακινήσεις και ε, δεν θα οδηγήσουν ποτέ στο να αντιμετωπίσουμε τις δευτερογενείς μετακινήσεις. Ο Άλτο Μόρο έλεγε ότι κανείς δεν μπορεί να επιλέξει να είναι στην Ευρώπη ή να είναι στην ε, Μεσόγειο, γιατί όλη η Ευρώπη είναι στη Μεσόγειο. Η αρχή αυτή πρέπει πάντα να είναι μπροστά μας, όχι μόνο για να αντιμετωπίζουμε τη σωστή προοπτική του ζητήματος τη μετανάστευσης. Πρέπει να είναι μπροστά μας και εκεί που διακυβεύεται η ίδια η ασφάλεια της Ευρώπης. Η υποστήριξη της ε, πολιτικής, των πολιτικών εξελίξεων στη Λιβύη ή ο ρόλος της Ευρώπης στη Μέση Ανατολή. Η Ιταλία τάσεται υπέρ του ρόλου μας και της δράσης μας στη Μεσόγειο. Επισκέφθηκα την Αλγερία και την Τινησία και είχαμε και τη διάσκεψη του Παλέρμου το Νοέμβριο πέρσι. Σύντομα θα επισκεφθώ το Μαρόκο. Πρόκειται για μια συνεκτική στρατηγική της Ιταλίας για να συνδράμουμε και εμείς στη σταθερότητα και σταθεροποίηση της κατάστασης, να αντιμετωπίσουμε τις αλλεπάλληλες κρίσεις προς συμφέρον όχι μόνο της χώρας μας, αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. Η Ευρώπη, πέρα από την Μεσόγειο, θα πρέπει να επενδύσει σε αυτή τη συνεργασία για την Αφρική και υπέρ της Αφρικής. Διαφορετικά, ε, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους επαναπατρισμούς που χρειάζονται μια συντονισμένη δράση της Ευρώπης αλλά και των κρατών μελών μεμονωμένα. Αυτό αφορά συγκεκριμένες απαντήσεις. Το μέλλον μας Αφρι... στην Αφρική πλαισιώνει αυτή την προσέγγιση. Και εγώ είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Γι' αυτό επισκέφθηκα τον Νίγηρα και το Τσάντ στα μέσα του Ιανουαρίου. Θα πρέπει λοιπόν μέσα στα πλαίσια των αξιών μας να προβούμε σε μία νέα προσέγγιση υπέρ της Αφρικής, ένα νέο μοντέλο συνεργασίας ως ίση μεταξύ ίσων, αναλαμβάνοντας αμοιβαία ευθύνες. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε αμέτωχοι στο γεγονός ότι ο πληθυσμός της Αφρικής, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες φτώχειας παρά τους φυσικούς πόρους που διαθέτουν αντιστοίχως. Ούτε μπορούμε να είμαστε αμέτωχοι στο γεγονός ότι η αφρικανική οικονομία χάνεται σε μερικές χιλιάδες υπεράκτιες επιχειρήσεις που επενδύουν σε φορολογικούς παραδείσους. Χαίρομαι γιατί η προτεραιότητα συνεργασίας με την Αφρική έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαριστώ τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ που έδωσε αυτή τη νέα όθηση για το κοινό μας μέλλον αναγνωρίζοντας αυτή την προτεραιότητα. Αυτό σημαίνει βέβαια και εγγραφή πιστώσεων καθώς και νέους τρόπους παρέμβασης. Η Ευρώπη θα πρέπει να ε, γράψει έναν απογραφικό κατάλογο βέλτιστων πρακτικών για να έχουμε μια ίση συνεργασία. Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό μέσα στα πλαίσια και του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 21-27. Η Ευρώπη θα πρέπει να έχει τα κατάλληλα μέσα και εργαλειοθήκες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεταναστευτικές ε, ροές, ιδιαίτερα στις ε, χώρες διαμετακόμισης. Και αυτό αφορά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Έξι δις ευρώ δόθηκαν στην Τουρκία για αυτό το σκοπό. Το Trust Fund υπέρ της Αφρικής έχει ένα κενό 550 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης έχει μεγάλη σημασία και η εσωτερική διαχείριση της μετανάστευσης. Δεν μπορούμε να μιλάμε για προστασία των παρακτήων μας ή την προστασία με βάση την σύνοριοφυλακή. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η πρώτη χώρα μετανάστευσης, αλλά και το ζήτημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί δραστικά. Οι μεταναστευτικές ροές δεν φτάνουν από μόνες τους. Έχουν κάποια αιτία, γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συλλογικά. Ο κανονισμός του Δουβλίνου του, που εγκρίθηκε το 2017, το Νοέμβριο του 2017, δεν επιλύει από μόνος του το ζήτημα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνδράμουν με αλληλεγγύη και υποχρεωτικά. Γι' αυτό στις 28 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μίλησε για την αρχή της αλληλεγγύης και της ίσης κατανομής αρμοδιοτήτων, καθώς και το άρθρο 80 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν βλέπουμε τις καταχρήσεις, το τι γίνεται με τις ανθρώπινες ζωές, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το δίκτυο των διακινητών που αποτελούν μεγάλη μάστιγα για την ανθρωπότητα και βεβαίως απειλή για την ασφάλειά μας. Ας μην είμαστε διχασμένοι, ας μην είμαστε ούτε ε, λαϊκιστές, αλλά ούτε υπέρ και της απόλυτης αποκέντρωσης. Σας έχουμε μία κοινή Ευρώπη, μία Ευρώπη της ενότητας και της ασφάλειας. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν δίχασμοι μεταξύ περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε και για την ΟΝΕ, την ολοκλήρωσή της, τη στιγμή που υπάρχουν εμπορικές και οικονομικές εντάσεις που κλειδονίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό αφορά και τα εθνικά χρέη ως ποσοστιαία αναλογία του ΑΕΠ. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μία επανισορρόπηση και επιμερισμός ευθυνών για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Δεν μπορεί να υπάρχει αυστηρή λιτότητα. Με βάση το δημοσιονομικό νόμο του 2019 από την Ιταλική κυβέρνηση πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε στις σωστές ε, αναθεωρήσεις και μεταρρυθμίσεις χωρίς να αποτελέσουν συσήφιο έργο. Έχουμε προωθήσει τη σταθερότητα και σταθεροποίησή μας μέσα στα πλαίσια του δημοσιονομικού εγχειρήματος και φυσικά η Ιταλική κυβέρνηση θα προωθήσει αυτή την πορεία. Παράλληλα, η προώθηση των δημοσίων επενδύσεων μέσα στα πλαίσια του ρυθμιστικού δικαιοδοτικού πλαισίου οδηγούν σε ένα σε μια δυναμικότητα της εθνικής μας ε, οικονομίας. Η οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να φτάσει σε μια εξισορρόπηση ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και το σχέδιο Juncker, το οποίο αποτελεί ευρωπαϊκή αναγνώριση της ανάγκης της δημόσιας παρέμβασης υπέρ των επενδύσεων. Τι σημαίνει να αντιμετωπίσουμε τη λιτότητα, όχι ότι δεν κατανοούμε την χρηματοοικονομική σταθερότητα, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική σταθερότητα και την αηφόρο ανάπτυξη. Ο Ζαν Κλοντ Ιούνκερ αναφέρθηκε στην ελληνική κρίση και το γεγονός ότι η λιτότητα ίσας ήταν υπερβολική και παρακινδυνευμένη. Γνωρίζω ότι μερικοί σε ορισμένα χρόνια θα ζητήσουν συγνώμη επίσης για την έλλειψη αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ή της κοινωνικής Ευρώπης. Ήδη Σήμερα θα πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες για την Ευρώπη του αύριο, ιδιαίτερα για τους νέους, για την εκπαίδευση, για τις καινοτομίες και για τις δημόσιες επενδύσεις που θα στρέφονται σε αυτούς τους στόχους. Γιατί μας ενδιαφέρει η αντιμετώπιση της, ε, του μεγαλύτερου ελλείμματος που υπάρχει. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική ενίσχυση και ανάπτυξη μετά από τη συνθήκη του Μάστριχτ και τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε να ε, διανύσουμε ακόμα πολύ δρόμο. Οι κρατικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει αυτή την πτυχή του ζητήματος. Το Eurogroup της 21ης Ιανουαρίου και η διάσκεψη κορυφής του Δεκεμβρίου όρισε μία ε, ομάδα υψηλών αξιωματούχων για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και το θέμα των τραπεζικών κλειδονισμών και της Τραπεζικής Ένωσης. Βεβαίως, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεθούν λύσεις σε υψηλό επίπεδο. Και η εξυγίαση των τραπεζών είναι ύψης της σημασίας. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν φτάσουμε σε μία νέα ύφεση, πριν φτάσουμε σε μία νέα παλινοδία. Με τη συνθήκη του Μάστριχτ ε, μιλάμε για την αντιμετώπιση των εθνικών χρεών, του εθνικού χρέους, σε σχέση 60% χρέος ΑΕΠ. Χρέος ΑΕΠ. Αυτό είναι το όριο και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η ΙΠΑ συνέδραμαν στην παγκόσμια οικονομική κρίση. Για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα πιο αποτελεσματικά, θα πρέπει να δημιουργηθούν κοινά μέσα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των κρίσεων συνδράμοντας με ευθύνη και αλληλεγγύη. Εάν δεν υπάρχει αρκετή αλληλεγγύη, μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί δεν έχουμε και μια κοινωνική Ευρώπη. Οφείλεται στην έλλειψη επαρκούς αλληλεγγύης. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατά προτεραιότητα την ανεργία και την υποστήριξη της ανάπτυξης. Να δοθεί μια όθηση σε αυτές τις προτεραιότητες με, τη, με συγκεκριμένα μέσα και εργαλειοθήκες για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Η διαφορά ανεργίας που πλήττει τους νέους που έχουν δυσθεώρητους δείκτες ανεργίας οδηγεί σε εθνικισμούς, σε εθνικιστικά στεγανά. Γιατί φυσικά οι χώρες που ευημερούν δεν θέλουν να αναλάβουν αυτό το κόστος, ενώ οι μειονεκτούσες περιφέρειες θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια αηφορίας μία πιο δίκαιη και πιο ίση Ευρώπη θα πρέπει να αφορά και το επόμενο πι μέσα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων. Να μην χάσουμε αυτή την προτεραιότητα. Με βάση και τις ε, υπαρξιακές μας προκλήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε την κατάλληλη εξισορρόπηση μεταξύ των νέων προτεραιοτήτων, μεταναστευτικό, ανάπτυξη, επενδύσεις, ασφάλεια και παραδοσιακές πολιτικές. Η ΚΑΠ θα πρέπει να τύχει της πλήρους υποστήριξής μας, καθώς και να προωθήσουμε την συνδρομή υπέρ μιας κοινωνικής Ευρώπης. Πολλές άλλες είναι οι προκλήσεις που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε να προωθήσουμε μια πιο, ένα πιο ίσο διεθνές εμπόριο υπέρ των καταναλωτών. Να προβάλλουμε κάθε πρωτοβουλία για να λάβουμε υπόψη και να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές και να συνδράμουμε στην προστασία των ηλικιωμένων και στην ψηφιακή εποχή, γιατί τα δικαιώματα ενέχουν και ένα κόστος. Η ε, Ευρώπη θα πρέπει να είναι ένα security provider, λαμβάνοντας υπόψη και τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, έχει μεγάλη σημασία το αρχικό μας μέλημα. Ποια Ευρώπη θέλουμε, ποια Ευρώπη χρειαζόμαστε, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορέσουν να συνεχίσουν να έχουν μία ειρήνη που διαρκεί ήδη 60 χρόνια. Η απάντησή μου είναι για άλλη μια φορά η ίδια. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι κοντά στους λαούς της. Η Ευρώπη του 21ου αιώνα θα πρέπει να συνεχίσει αυτό το σχέδιο υπέρ των λαών, με τους λαούς, για τους λαούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυτό το συγκεκριμένο ρόλο ενίσχυσης του νομοθετικού έργου γιατί έχετε εκλεγεί με καθολική ψηφοφορία, εκπροσωπείτε άμεσα τον Ευρωπαίο πολίτη και φυσικά υπάρχει και το θέμα λογοδοσίας έναντι των άλλων θεσμικών οργάνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ανταποκριθεί στις αλλαγές, αλλαγές ιστορικής σημασίας που άλλαξαν τα γεωπολιτικά δεδομένα. Παράλληλα, χρειάζεται μία ενίσχυση της άμεσης δημοκρατίας έτσι ώστε να ανακτήσουμε την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων έναντι των πολιτών. Το ευρωπαϊκό σενάριο ορίζει ορίζει και ορίζεται από την απογοήτευση των πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε την στάση των πολιτών και αυτό αφορά και την Ιταλία που πολλές φορές δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς. Χρειάζεται αυτή η αλλαγή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σωστή εκπροσώπηση θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή αυτές τις αρχές. Σας δούμε το Brexit, θέμα ύψης της σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα προσεχή χρόνια. Μπροστά σε αυτή την ε, πρόκληση η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ενωμένη και αλληλέγγυα. Μετά από 60 χρόνια ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης χωρίς να υπάρχουν ε, κυρωτικού τύπου αντιδράσεις. Πρόκειται για μία περίοδο χωρίς προηγούμενο. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες και τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό που θα ανακύψει μετά από το Brexit. Κύριε Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να δούμε τι δεν λειτουργήσε σωστά και μέσα από τις συνθήκες και να αποφύγουμε τις φυγόκεντρες ε, δυνάμεις, όπως ισχύει και στη χώρα μου και είναι απότοκο της απογοήτευσης των πολιτών. Εάν θέλουμε η Ευρώπη να είναι το κοινό μας μέλλον, θα πρέπει να περάσουμε από το λόγο στην πράξη. Να ορίσουμε μια νέα Ευρώπη την Ευρώπη των λαών πιο αλληλέγγυα, πιο ίση, πιο δίκαιη, πιο δημοκρατική. Τη μοναδική όπου οι πολίτες σήμερα και αύριο θα αξίσει να ζουν για αυτήν και μέσα από αυτήν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ. Πριν δώσω το λόγο στον αντιπρόεδρο της Επιτροπής κύριο Κατάινεν να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι για μας να μετέχουν τα κράτη-μέλη στις ε, προσπάθειες ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση ζητούμε μια μεγαλύτερη δέσμευση στις επόμενες συνεδριάσεις του Συμβουλίου ούτω ώστε να γίνουν δεκτές οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ενδεχόμενα κάποια, κάποιο συμβασμό για τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου. Νομίζω ότι αυτά που λέω αντικατοπτρίζουν τι απόψει όλων ε, στο, στο, στην Ολομέλεια. Ο κύριος Κατάινεν έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε Ταγιάννη, κύριε Πρωθυπουργέ Ταγιάννη, αξιότιμα μέλη. Η Ιταλία φυσικά ε, κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της Ευρώπης. Έχει δώσει τόσο πολλά στην Ευρώπη. Είναι ιδρυτικό μέλος από την αρχή διαμόρφωσε την Ένωσή μας ε, σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Οι Σπινέλοι εν Ρώση είχαν ε, κρατούντο σε ένα νησί της Ιταλίας και εκεί εξεπώνησαν ένα σχέδιο για μια ελεύθερη και ενωμένη Ευρώπη. Κάλεσαν τα έθνη της Ευρώπης που τότε ήταν ε, αντιμέτωπα να συμμαχίσουν ούτως ώστε τα σφάλματα του παρελθόντος να μην επαναληφθούν. Μετά τον πόλεμο. Ο Ντεγκάσπερη έγινε ένας από τους ιδρυτικούς πατέρες της Ευρώπης. Και το 1957 στο Καπιτόλιο, στον λόφο του Καπιτολίου υπεγράφει η Συνθήκη της Ρώμης και δημιουργήθηκε η Ένωσή μας με έξι ιδρυτικά κράτη-μέλη. 60 χρόνια κατόπιν, το 2017, άλλη μια φορά, σε αυτά τα ίδια σκαλοπάτια της ε, Ρώμης, οι ηγέτες των κρατών μας στάθηκαν ο ένα δίπλα στον άλλον για να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για την Ένωση. Αυτή τη φορά ήταν 27 από όλες τις γωνιέ της Υπήρου μα. Αυτό είναι δείγμα του πόση πορεία έχουμε διανύσει. Το τονίζω αυτό γιατί η ειδική ιστορία της Ιταλίας είναι ένας από τους πολλούς λόγους που έχει μία τόσο μοναδική και σημαντική θέση στην Ένωσή μα. Αλλά επίση, γιατί καταδεικνύει ότι η Ευρώπη προοδεύει, ότι η Ευρώπη επιτυχάνει τα μεγαλύτερα επιτεύγματά της όταν ε, έχει την Ιταλία και τους Ιταλούς ως παλόμενη καρδιά της. Η ιστορία αυτή πρέπει να μας βοηθήσει να είναι οδηγός και για το μέλλον. Για να υπάρξει ένα επιτυχές μέλλον για την Ένωσή μας, η Ένωση χρειάζεται στην καρδιά της μια ισχυρή Ιταλία. Μια Ιταλία, από την άλλη μια χρειάζεται μια ισχυρή και πρωτοπόρα Ευρώπη. Πρέπει να οικοδομήσουμε από κοινού το κοινό μας μέλλον. Ενωμένοι, και με αλληλεγγύη. Συνεργαζόμενοι πάντα και όχι αντιπαρατηθέμενοι. Συζητώντας και όχι ο καθένας για τον άλλον, σχολιάζοντας τον άλλον. Και αν θέλουμε να έχουμε μια πραγματική ένωση αλληλεγγύης, η Ιταλία είναι το καλύτερο μέρος για να ξεκινήσουμε. Εκεί ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για να βοηθήσει την Ιταλία να ε, ανοικοδομηθεί μετά τους τρομερούς σεισμούς του 1960. Κινητοποιήθηκαν πολλές χιλιάδες νέοι και εδόθησαν και 1,2 δισεκατομμύρια με βάση τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης. Όλοι είδαμε τις εικόνες αυτών των νέων εθελοντών από όλα τα μέρη της Ευρώπης που βοήθησαν να ξαναχτιστεί η αρχαία και πανέμορφη εκκλησία της Νόρσια. Αυτή είναι η αλληλεγγύη η οποία είναι η βάση της ενωσής μας και πρέπει να συνεχίσει να είναι η βάση του κοινού μας εγχειρήματο. Η Ιταλία επέδειξε το ίδιο πνεύμα. Αμέτρητες φορές όλα αυτά τα χρόνια. Ο, πρόεδρο πρόεδρος Γιούνκερ το έχει πει επανειλημμένα. Η Ιταλία είναι ε, μία από τις χώρες που έσωσαν την τιμή της Ευρώπης ε, στην κορύφωση της ε, κρίσης ε, των προσφύγων. Γιατί ορισμένοι βραδιπόρησαν να στηρίξουν τις προσπάθειες της Ιταλίας. Αλλά επίσης είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη στο μεγαλύτερο μέρος της στήριξε όσο μπορούσε την Ιταλία. Από τότε που ξεκίνησε η μεταναστευτική κρίση μέχρι το τέλος του 2018 η Επιτροπή διέθεσε σχεδόν 950 εκατομμύρια για να στηρίξει τις ε, πολιτικές αυτές στην Ιταλία. 225 εκατομμύρια συγκεκριμένα δόθηκαν για επίγουσα βοήθεια για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης και να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις υποδοχής και να στηρίξει όλες τις αρχές και ε, τους πολίτες που βοηθούσαν. Η Ευρώπη στάθηκε στο πλευρό της Ιταλίας. Και να μην ξεχνάμε την επιχείρηση Σοφία ή το ρόλο της Ευρωπαϊκής Άκτο και Σύνορο Φυλακής που σώζει ζωές στη θάλασσα. Αυτό είναι μια κοινή προσπάθεια και γι' αυτό χρειαζόμαστε την Ιταλία. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να υπερβεί τις διαφορές της για να καταλήξει σε βιώσιμες και υπεύθυνε λύσεις. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να στηριζόμεθα σε ad hoc λύσεις. Βεβαίως έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που είχαμε την ε, κορύφωση, την κορύφωση της κρίσης όπου 80% ε, των ε, προσφύγων έφταναν ε, στην κεντρική Μεσόγειο. 7.000 ζωές σώθηκαν στη θάλασσα. Αλλά τώρα πρέπει να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια αυτή, να κάνουμε τις αναγκαίες αλλαγές στο σύστημα ασύλου μας. Η Επιτροπή έχει υποβάλει πολλές προτάσεις και τώρα πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να συμμετάσχει πλήρως η Ιταλία αν θέλουμε να επιτύχουμε σε αυτό το εγχείρημα. Αξιότιμα μέλη, κύριε Πρωθυπουργέ, Ευρώπη σημαίνει ειρήνη και ευημερία. Και είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την υπεράσπιση των αξιών της. Όλοι μαζί. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να επιτύχει η Ευρώπη.